Η περίοδος συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διακόπηκε στις 14 Απριλίου συνεχίζεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι περισσότεροι ξέρουν ακριβώς τι έγινε στις 29 ε, Απριλίου 1986